Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω λάβει τις εξής υποψηφιότητες. Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο, Κορίνα Κρέτσου, Ρίχαρτ Τσανέτσκι, Ινδικο Γκάλ Πέλτς, Σιλβί Αλεξάνδρ Γκραφ Λάμστορ. Ουλρίκε Λούνατσεκ. Μέριτ Μαγκίνε. κ. Δημήτρη Παπαδημούλης. Όλη Ρεν. Νταβίτ Μαρία Σασόλη. Αντώνιο Ταγιάννη. Ραμόν Λουίς Βαλκάρσελ Σισό. Αντίνα Ιωάννα Βαλεάν και Ράινερ Βίλαντ. Οι υποψήφοι και υποψήφιες μου διαβίβασαν ότι συμφωνούν με ε, την υποβολή αυτή των υποψηφιωτήτων. Ερχόμαστε στην εκλογή αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να ορίσουμε δύο ακόμη ψηφολέκτες διότι απουσιάζουν δύο συνάδελφοι που ήταν ψηφολέκτες το πρωί. Λοιπόν, σαν νεράιδα τώρα εγώ, θα τραβήξω δύο ονόματα. Όλε Λούτβιξον. Όλε Λούτβιξον. Όλε. Όλε. Peter Lundgren. Και ο Peter Είναι παρόν ο κύριος Λούντκρεν. Μάλιστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Also, Herr Λοιπόν, ο κύριος Λούντβιξον και ο κύριος Λούντκρεν ορίζονται νέοι ψηφοδελέκτες ε, ε με G, κύριε Λουτβιξόν, στην κάλπη αυτή και ο κύριος Λούντκεν στην κάλπη H μέχρι K. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων είναι ε, μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων στο Προεδρείο. Χρειάζεται μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού. Θα σας διαβάσω μία φορά το άρθρο αυτό για να καταλάβουμε τι κάνουμε και μετά θα σας εξηγήσω οι αντιπρόεδροι εκλέγονται ε, σε ένα ψηφοδέλτιο και ε, μέχρι 14 αν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία με τη σειρά ε, των ψήφων που έλαβαν θεωρούνται ότι εκλέγονται. Αν μετά δεν έχει καλυφθεί ο αριθμός, είναι μικρότερος από τον προσφλήρωση εδρών, διεξάγεται και δεύτερη ψηφοφορία με τους ίδιους όρους για να πληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες αν απαιτηθεί και τρίτη ψηφοφορία, τότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλεγέντες θεωρούνται οι πρεσβύτεροι από τους υποψηφίους. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια έχουν διανεμηθεί και τώρα παρακαλείστε να τα χρησιμοποιήσετε. Παρακαλώ βάλτε σταυρό στο κουτάκι δίπλα ε, στο όνομα του υποψηφίου της υποψηφίας της αρισκίας σας και θέλω να σας δώσω την εξής ε, συμβολή. Είναι 14 οι αντιπρόεδροι που πρέπει να εκλεγούν και μπορείτε να βάλετε μέχρι και 14 σταυρούς. Αν βάλετε παραπάνω είναι άκυρα μπορείτε από ένα σταυρό να βάλετε ή σε ένα όνομα ε, που θέλετε, αλλά μέχρι 14. Πάνω από 14 θα θεωρηθεί άκυρο το ψηφοδέλτιο. Ich den zwar noch nicht eröffnet, aber mir... Δεν είπα ότι άρχεται η ψηφοφορία, αλλά μα θέλετε να ορμήσετε παρακαλώ, τι να πω. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. Κύριε Γκίλ, θέλετε το λόγο. Ορίστε. Das ist jetzt sinnlos. Thank you, President. I was trying to get attention. Ευχαριστώ. Προσπαθούσα να τραβήξω την προσοχή σας ε, νωρίτερα, διότι δυνάμει του άρθρου 17 δεν αποκλείεται να ακούσουμε τους ε, ε, υποψηφίους ε, για τη θέση αντιπροεδρού όπως έγινε με τους υποψηφίους για την προεδρία. Δεν χρειάζεται να μιλήσουν τόσο πολύ. Ένα λεπτό έκαστος ήταν αρκετό για να σχηματίσουμε και μια εικόνα για ποιον ψηφίζουμε. νομίζω ότι θα βοηθούσε αυτό για λόγους διαφάνειας διότι είναι πολύ άριθμα τα νέα, οι νέοι βουλευτές. Ναι, όπως βλέπετε κύριε Αγγέλη, τώρα αυτό το θέμα έχει λήξει, είναι θεωρητικό μάλλον και δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε επί της ουσίας. Οι συνάδελφοι ε, είχαν τέτοια λαχτάρα να ψηφίσουν που δεν περίμεναν να πω ότι αρχίζει η ψηφοφορία καν. Που δείχνει ότι η δημοκρατία δημιουργεί τη ζωή της, τη φτιάχνει μόνη της. Ε, έχετε δίκιο, αλλά τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ αυτό. Haben alle Abgeordneten ihre... Ψηφίσανε όλοι οι βουλευτές παρακαλώ. Ah, ja. Okay. Ja, ja, ja. Il y a encore des filles. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, εψήφισαν όλοι οι βουλευτές, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει. meine... Κυρίες και κύριοι, ρωτώ για τελευταία φορά. Εψήφισαν όλοι οι βουλευτές, παρακαλώ. Ωραία. Εψήφισαν και οι ψηφολέκτες. Ψήφισαν και οι ψηφολέκτες, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Ωραία. Λήξεις της ψηφοφορίας. Παρακαλώ τους ψηφολέκτες να μεταβούν στην αίθουσα R11 για να προχωρήσουν στην καταμέτρηση. Διακόπτε τη συνεδρίαση. Θα ακούσετε από το κουδούνι πότε θα επαναληφθεί και θα δείτε και στις οθόνες ε, την ώρα επανέναρξη. Διακοπή λοιπόν τη συνεδρίαση.